Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση. Έκθεση Μάντερς, ονομασίες και επισήμανση κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Δίνουμε τον λόγο στον κύριο Μάντερς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίσατε γρήγορα, και δεν ήμουν προετοιμασμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες για την καλή συνεργασία που είχαμε με όλους τους σκιώδεις ηγητές. Να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο γιατί χάρη στην Ουγγρική Προεδρία θεωρώ πως ε, ε, καταφέραμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα εδώ πέρα. Πρόκειται περί ενός κανονισμού εδώ πέρα και όχι οδηγίας γιατί εγώ θεωρώ πως ε, καλύτερο είναι οι κανονισμοί σιγά σιγά να επικρατήσουν όπως πρότεινε και ο καθηγητής ο κύριος Μόντι στην έκθεσή του γιατί κάνουμε πάρα πολλά νομοθετήματα τα οποία εφαρμόζονται διαφορετικά και άρα ε, έχουμε βελτιώσει κάποια πράγματα. Η πρόταση της ε, Κομισιόν βελτιώνει την ε, προστασία των καταναλωτών καθώς στην αρχική πρόταση δεν αναφέρονταν σχεδόν καθόλου οι καταναλωτές και θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν υπόψη στην έκθεση αυτή κάτι το οποίο έκανα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημεία τα οποία είναι σημαντικά εδώ πέρα δηλαδή ε, μια έρευνα για τις αλλεργικές αντιδράσεις. Η Κομισιόν είπε πως ε, δέχεται να κάνει κάτι τέτοιο και άρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 θα παρουσιαστεί η σχετική ε, μελέτη και τα αποτελέσματα αυτά θα πάνε σε μια κάποια νομοθεσία και έχει δηλώσει το Συμβούλιο πως θα ε, τα εξετάσει. Επίσης ε, αντιδράσεις ε, αλλεργικές σε χημικές ουσίες καθώς ξέρουμε πως πάρα πολλοί καταναλωτές έχουν πλέον τέτοιες αντιδράσεις και θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη προειδοποίηση. Επίσης συχνά υπάρχουν παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, αλλά βλέπετε πως ε, όσον αφορά την ε, προέλευση των προϊόντων και το λεγόμενο made in ε, δεν σημαίνει αυτό καθόλου αυτό το οποίο φαντάζεται ο καταναλωτής οπότε ζητάμε από την Κομισιόν να ερευνήσει εάν είναι δυνατόν να καταστεί σαφές πως εάν ε, ένας κατασκευαστής λέει πως κάτι έχει φτιαχτεί στην Ολλανδία ή στην Ιταλία να έχει πραγματικά παραχθεί εκεί πέρα και όχι να είναι 99% στην Κίνα και βάζουν ένα κουμπάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λένε ότι έχει φτιαχτεί στην Ευρώπη. Επίσης, αντιγραφές. Κοιτάξτε, ε, θα μπορέσουμε να δούμε, να ερευνήσουμε αν μπορούμε να έχουμε όχι μόνο μία απλή φασμάτινη ετικέτα, αλλά να ενημερώσουμε με βέλτιστο τρόπο τον ε, καταναλωτή με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Επίσης, ε, δέχτηκε το Συμβούλιο να υπάρχει δήλωση του εάν υπάρχουν ζωικά προϊόντα στα ενδύματα, καθώς είναι δύσκολο να ξεχωρίσει ο καταναλωτής εάν είναι γούνινο ή απομίμηση γούνας και είναι σημαντικό αυτό για πολλούς ε, καταναλωτές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί καθώς ε, σιγά σιγά υπάρχει η επικράτησή του θα πρέπει να υπάρχουν και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη σχετική σήμανση. Επίσης δεν είναι ανάγκη στο σύγχρονο κόσμο να έχουμε 23 γλώσσες στην ε, ετικέτα. Θεωρώ πως ε, η δήλωση του Συμβουλίου θα δημιουργήσει αρκετή νομίζω εμπιστοσύνη στους ε, καταναλωτές και ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου για το καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε κύριε Μάντερς για το Συμβούλιο κυρία Κιόρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιγητά, κύριε Επίτροπε, κυρίες ε, και κύριοι. Είναι θετικό το ότι είχαμε συμφωνία στην δεύτερη ανάγνωση για πρόταση κανονισμού για την σήμανση κλωστοϊφατουργικών προϊόντων. Τώρα λοιπόν έχουμε το αποτέλεσμα των τριών αυτών οδηγιών που καταργήθηκαν. Πράγματι, συμφωνώ και εγώ, ήταν πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Οφείλουμε να ευχαριστούμε τον κύριο Τόινε, οφείλουμε τον κύριο για την καλή συνεργασία στην διαδικασία αυτή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Σουηδική, Ισπανική και Βελγική Προεδρία γιατί το αποτέλεσμα αυτό δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τις ε, δικές τους εργασίες. Η ΔΕ Κομισιόν έπαιξε επικοδομητικό ρόλο σε όλη την ε, διάρκεια αυτού του εγχειρήματο και αν όλα πάνε καλά το φθινόπωρο θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την ε, νομοθεσία αυτή η οποία θα ισχύσει από το 2012 και άρα συνεισφέρουμε έτσι τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού στο σημαντικό αυτόν τομέα. Οι υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις για χρήση κλώσεων προϊόντων ε, θα προωθήσουν την καινοτομία στον ε, κλάδο αυτών και έτσι θα έχουν οι καταναλωτές τα πλεονεκτήματα καινοτόμων προϊόντων. Η Ουγγρική Προεδρία είναι πεπισμένη πως ο κανονισμός θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και θα βελτιώσει την προστασία των ε, καταναλωτών. Επίσης θα υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης και άρα οι συνομοθέτες θα μπορέσουν να λάβουν υπόψη τις μελλοντικέ εξελίξεις γιατί η Κομισιόν θα υποβάλει και μια μελέτη για περαιτέρω απαιτήσει σήμανσης όπως παραδείγματο χάρη οδηγίες χρήσης, απλοποίηση των μεγάλων ε, ενδείξεων ε, σε ηλεκτρονική ετικετοθεσία, αλλεργικέ αντιδράσεις και άλλη τεχνολογία. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο τονίζουν πως ε, θα πρέπει να υπάρχει, να αποδείτε μεγάλη σημασία στην διχνηλασιμότητα των προϊόντων αυτών. Η δε νομοθεσία αυτή θα δώσει δυνατότητα γρήγορη γρήγορης αδειοδότηση αυτών των προϊόντων και θεωρούμε πως ε, θα υπάρξει και μια νέα απέτηση, δηλαδή να υπάρχει ένδειξη για ζωικά προϊόντα, για τις σύνες εκείνες οι οποίες είναι ζωικά προϊόντα. Επίσης ενισχύεται η νομική ασφάλεια γιατί μιλάμε περί κανονισμού και όχι οδηγίες. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Αγγιέρη ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Σταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μάντερς, τον εισηγητή δηλαδή, για τη δουλειά που έκανε, <laughs> μαζί με όλους τους υπολείπους συναδέλφου, με την Επιτροπή, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μετά από κάποιες διαπραγματεύσει που δεν ήταν καθόλου απλές και εύκολες. Θα, ε, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε μέσα στα πλαίσια της δεύτερης ανάγνωσης να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες μας, οι καταναλωτές μα, η βιομηχανία μα θα μπορέσει να αποφεληθεί από νέε ίνε, από καινοτόμα προϊόντα ε, τα οποία θα παράγουμε και θα επιτρέψουμε στις, ε, να μειωθεί το κόστος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το Κοινοβούλιο, το οποίο συμμετείχε σε αυτή την διαθεσμική συζήτηση με τις τροπολογίες τις οποίες υπέβαλε. Κάποιες από αυτές ε, τόνισαν ιδιαίτερα την πολιτική διάσταση και, το, και τα ενδιαφέρον των καταναλωτών για το θέμα αυτό. Στην πρώτη ανάγνωση που έγινε δεκτή από το Κοινοβούλιο τονίστηκε το, ότι θα, το γεγονός ότι θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την σήμανση των χριστιανικών προϊόντων και για την ετικέτα προέλευσης για πολλά προϊόντα. Ε, ξέρετε ότι μέσα στα πλαίσια των ζητήσεων στο Συμβούλιο ζητήθηκε να είμαστε πιο ευέλικτοι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ανάμεσα στα, στα θεσμικά όργανα. Το κείμενο που έχουμε στη διάθεσή μας αποτελεί ε, τον καρπό μιας συμβιβαστικής ε, λύσης, ε, πολύ ισορροπημένης, και ελπίζουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες ε, πρόοδοι, όπως είπε και η κυρία Γκιώρη στην ομιλία της. Ο καταναλωτής με τον τρόπο αυτό θα έχει περισσότερες πληροφορίες ε, όσον αφορά την, ε, τις σύνες που θα προέρχονται από ζωικά προϊόντα στο ύφασμα και θα ε, αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα κλουστοφορικά προϊόντα. Ένα άλλο στοιχείο είναι η απλούστευση. Η Επιτροπή θα αντικαταστήσει με τις ευρωπαϊκές, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ένα τεχνικό παράρτημα πάνω από 50 σελίδες. Όμως ε, υπάρχουν και άμεσα αποτελέσματα από αυτόν τον παρόντα κανονισμό που δεν αποτελούν όμως την τελευταία φάση της διαδικασίας. Αντίθετα είναι ένα σημείο εκκίνησης, μια αφετηρία για να συνεχίσουμε την ανάλυση και να βελτιώσουμε την, ε, το νομοθετικό κείμενο. Το κείμενο του νέου κανονισμού προβλέπει μια ρήτρα σφαιρικής αναθεώρησης που καλεί την Κομισιό να προβλέψει ε, και άλλες υποχρεώσεις, αν χρειάζεται δηλαδή, στον τομέα αυτό και η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις ε, για τους τομείς που απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση. Και εγώ αναλαμβάνω τη δέσμευση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασχοληθώ με αυτή την αναθεώρηση άμεσα και ενδελεχώς. Και είμαστε, έχουμε ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με τους καταναλωτές για πολύ βασικά θέματα. Τώρα ποιες είναι αυτές οι βασικές πληροφορίες και ε, πώς θα είναι αυτές οι βασικές πληροφορίες διαθέσιμες, πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις, ε, το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζουν την απόκτηση κλωστοβιτουργικών προϊόντων, πως ε, οι απαιτήσει βιωσιμότητας και ανιχνευσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης των εταιριών επηρεάζουν την αγορά των κλωστοφαντουργικών. Πώς ε, μπορούμε να, βελτι... να υποφεληθούμε περισσότερο από την τεχνολογία και πώς μπορούμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμόσουμε τις ε, τις νομοθετικές μας αριθμίσεις, ε, σεβόμενοι τις ε, κοινωνικές, ε, περιβαλλοντικές και οικονομικές απαιτήσεις. Αυτά είναι μια προκαταρκτική δουλειά κύριε, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα το θέμα της προέλευσης, το σήμα προέλευσης θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της, των εργασιών μας. Και με η επανεξέταση θα, επιτρέψει, θα μου επιτρέψει μάλλον να εκφράσω την υποστήριξή μου στο σήμα προέλευσης και θα χρησιμοποιήσουμε το Made In που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών θα τα εξετάσουμε τα θέματα αυτά πάρα πολύ προσεκτικά για να έχουμε σαφείς κανόνες, για να έχουμε σαφείς πληροφορίες και για να σεβαστούμε τις ευθύνε μας απέναντι στους καταναλωτές τη στιγμή που αγοράζουν τα προϊόντα. Η Κομισιόν θα εξετάσει επίσης και την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις αλλεργίες και στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τα κλεισιδωρικά προϊόντα. Θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση στον τομέα αυτό έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο, τρόπο την, την νομοθεσία που υπάρχει Παραδείγματο χάρη, με το made in, με το σήμα προέλευση, ο καταναλωτή θα είναι σίγουρο ότι αγοράζει ένα προϊόν, ένα ύφασμα, το οποίο δεν απειλεί την υγεία τη δική του των παιδιών του. Διότι ε, θα είναι σίγουρο ότι αγοράζει ένα προϊόν το οποίο αποτέλεσε καρπό θυσιών που, έχουν κάνει, που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο για άλλη μια φορά γιατί ε, υπογράμμισε τη σημασία αυτή την, ε, αυτής της ρήτρας, δηλαδή να συνεργαστούμε άμεσα με την Κομισιό για να προχωρήσουμε τον κανονισμό αυτό και θα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 θα υποβάλουμε μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Και εγώ θέλω να ε, περιορίσουμε τις προθεσμίες έτσι ώστε να υποβάλουμε την, το κείμενο αυτό να τον πιο γρήγορα και θα συστήσω στις, επιτρο... στις υπηρεσίες μου να επιταχύνουν τις εργασίες τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους ομιλητές των ομάδων. Πρώτα απ' όλα, κόμι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία σε αυτό τόσο σημαντικό θέμα και καταβάλαμε όλοι μια σημαντική προσπάθεια για να βρούμε ένα σημείο συνάντηση ανάμεσα στι ε, ε, συγκρουόμενε απόψει του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο στόχο μου ήταν, είναι και θα είναι να υιοθετηθούν δεσμευτικέ ε, ρήτρε όσον αφορά την σήμαση των κρυστανερικών προϊόντων. Ο καταναλωτή και οι εταιρείε πρέπει να προστατευτούν. Πιστεύω ότι ο συμβασμό στον οποίο καταλήξαμε σήμερα είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ζήτησα από του συναδέλφου μου να πολεμήσουν με το Συμβούλιο και δεν χρησιμοποιώ τον ε, όρο πολεμό, έτσι εύκολα. Ήταν δύσκολες οι συζητήσεις και το made in είναι πάρα πολύ σημαντικό και, το, και η ανεχνευσιμότητα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα ο Ευρωπαίος καταναλωτής βρίσκει στην αγορά κλωστοβερικά προϊόντα με το made in Italy, made in Germany, made in France ενώ η παραγωγή τους έγινε σχεδόν ολοκληρωτικά αλλού και θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες με το microchip και το RFID για την ε, σήμανση των προστατευτικών ε, προϊόντων έτσι ώστε να πατάξουμε την ε, παραποίηση. Πιστεύουμε ότι ο τομέας αυτός χρειάζεται στο άμεσο μέλλον προστασία και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την σημασία της ανιχνευσιμότητας και της προέλευσης και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον. Περιμένουμε βέβαια με μεγάλη ανυπομονησία την μελέτη που θα εκπονήσει η Κομισιόν και την ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και τον Επίτροπο ε, για την δέσμευση που ανάλαβε να ε, επισπεύσει τις προθεσμίες γιατί ο κλεισματουργικός τομέας χρειάζεται προστασία. Θα πρέπει οι πολίτες μας, οι καταναλωτές μας να έχουν μια ουσιαστική και πραγματική ενημέρωση αναφορά το προϊόν που αγοράζουμε και νομίζω ότι όλοι όλοι, ότι αυτή η απέτηση είναι προς το συμφέρον όλων μας, διότι όλοι είμαστε καταναλωτές. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά, η κυρία Σάλτε Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πολύ καλή συμβεβαστική λύση ε, που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον εισηγητή κύριο Μάντερς, ο οποίος ε, πρόθεσε ένα πνεύμα συνεργασίας πολύ καλό, πολύ θετικό στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε μια τεχνική πρόταση πριν από κάποιο καιρό, μια πρόταση η οποία είχε πλονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και μόνο. Μέσω όμως της κοινοβουλευτικής διαδικασίας καταφέραμε ευτυχώς ε, να προσθέσουμε στην πρόταση αυτή στοιχεία που πλέον ε, έχουν ως αποτέλεσμα το νομοθέτημα αυτό να είναι προς όφελος και των καταναλωτών. Έχουμε λοιπόν καλύτερη σήμανση και μεγαλύτερη ασφάλεια για τους καταναλωτές. Αν βέβαια υλοποιηθεί και εφόσον υλοποιηθεί αυτή η νομοθεσία, που είναι και το σημαντικότερο για μένα και την ομάδα μου αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μην υπάρχουν προβλήματα υγείας από να οφείλονται σε υφάσματα, σε κλωστοφαντουργικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ε, μόλις είπε και ο Επίτροπος, ε, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν ίχνη επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα τα οποία να προκαλούν αλλεργίες. Ε, μας ικανοποιεί η πρόταση αυτή. Επίσης ε, η συμφωνία για την προέλευση και την ανιχνησιμότητα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο για τους καταναλωτές, είναι κάτι που το επιθυμούν. Και εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα να πάμε λίγο πιο πέρα, να εναρμονίσουμε τα μεγέθη ε, των ρούχων, να εισαγάγουμε νέε τεχνολογίες στη σήμανση των κλωστοφαντουργικών προϊόντων στο μέλλον και ούτω καθεξής. Πάντω, πρόοδο επιτελέστηκε και πρέπει να μάθουμε και το εξή ότι η νομοθεσία που προτείνουμε πρέπει να είναι προ όφελο και των επιχειρήσεων αλλά και των καταναλωτών. Αυτό είναι ο καλύτερο δυνατό τρόπο να έχουμε μια εύρυθμη αγορά εσωτερική. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου ε, για το πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Σάλτε Μόσε. Για ένα μισή λεπτό, κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόιν Μάντερς για την επιμονή που έδειξε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Καλωσορίζω τη συμφωνία που επιτεύχθη στη δεύτερη ανάγνωση. Αν και μπορεί να βελτιωθεί, παρόλα αυτά θα επιφέρει καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών. Υπάρχουν πολλές θετικές στοιχές. Πρώτα απ' όλα η διαδικασία που απλοποιεί το παράρτημα 1 θα μειωθεί έτσι το διοικητικό κόστος για την κλωστοϊφαντουργία και θα μπορέσει να πάει ε, τα κονδύλια αυτά να πάνε στην καινοτομία και άρα είναι αυτό υποφελές για τους καταναλωτές. Θεωρώ πως ο οργανισμός αυτός έχει πλέον εκτήματα για τους καταναλωτές λόγω των απαιτήσεων σήμανσης. Οι επαρκείς πληροφορίες για τα προϊόντα πριν αγοραστούν αυτά είναι κάτι το φυσικό. Οι συζητήσεις για τη σήμανση ήταν μακροσκελέστερες από τις συνήθως, αλλά αυτό μόνο θα ωφελήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Χρειαζόμαστε πράγματι περισσότερο χρόνο για να δούμε τον αντίκτυπο που έχουν περαιτέρω απαιτήσει ε, σήμανσης. Γι' αυτό είναι ένα πρώτο βήμα η μελέτη της ε, Κομισιόν. Και επίσης ε, σημαντικό είναι η σήμανση ζωικών υλικών γιατί κάποιοι καταναλωτές δεν θέλουν να αγοράζουν τέτοια προϊόντα. Συνολικά λοιπόν θα ε, βοηθήσει την εσωτερική αγορά και υποστηρίζω αυτή την, ε, τον κανονισμό. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά. Ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ. Η απλούστευση των κανονισμών και των ρυθμίσεων που αφορούν ε, την σήμανση των κλωστοφαντουργικών προϊόντων έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων ε, υφάνσιμων ινών και την εισαγωγή τους στην αγορά. Η πρόταση που θα ψηφίσουμε αύριο ε, διαφέρει κατά πολύ από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ουσιαστικά εισήγαγε τεχνικές τροποποίησεις και ρυθμίσεις. Ο γενικός στόχος πλέον είναι να επιταχυνθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και καταχώρησης νέων υφάνσιμων ινών που χρησιμοποιούνται στην κλωστεφαντουργία. Ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται όμως ότι θα μπορούν τα νέα προϊόντα, οι νέες ίνες να χρησιμοποιούνται πιο γρήγορα από τους καταναλωτές. Οι εργασίες που έγιναν οδήγησαν σε πολύ σημαντική απλούστευση των διαδικασιών. Επίσης, το Κοινοβούλιο πρότεινε να ε, υπάρξει σημαντική βελτίωση στους κανόνες περί προέλευσης και χώρων προέλευσης. Είναι θετική η συμβιβαστική λύση που επιτεύχθη, αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα μου είχε ζητήσει να γίνει δεκτή η αρχική πρόταση της Κομισιόν, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορα πλεονεκτήματα και ωφέλη και για τους επιχειρηματίες της αγορές και για τους καταναλωτές. Η Κομισιόν θα πρέπει να κληθεί να αναλύσει σε μεγαλύτερο βάθος ε, τη σήμανση των κλωστοδουρικών ε, προϊόντων που παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέχρι, ε, το 2013 θα πρέπει να δημοσιοποιήσει μια έκθεση σε σχέση με το νέο σύστημα σήμανσης ε, των κλωστοδουρικών προϊόντων που θα συνοδεύεται ίσως και από μια νέα νομοθετική πρόταση. Ελπίζουμε να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Αν συνεχίσουμε να παρέχουμε καλή ενημέρωση στους καταναλωτές και αν συνεχίσουμε και το δικό μας έργο σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση, την εναρμόνιση των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϊφαντουργία, θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη μας τους στόχους τη της προστασίας των καταναλωτών αλλά και των ωφελών για τη βιομηχανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σβένσον για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντα λέμε πως είναι σημαντικό να έχει δύναμη ο καταναλωτής. Εάν τα εννοούμε αυτά, πρέπει να κάνουμε και κάτι ανάλογο και να δώσουμε στους καταναλωτές αυτή τη δύναμη. Να έχουν δηλαδή αρκετές πληροφορίες για τα προϊόντα για να μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις τους. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Στάντερς για την επιμονή του για το ότι διασφάλισε πως τα ζητήματα των καταναλωτών περιέχονται εδώ πέρα. Επίσης για το ότι έδειξε τόσο μεγάλη διάθεση να αυξηθεί η δύναμη των καταναλωτών. Έχω καταθέσει τροπολογίες εξ ονόματος του για την προέλευση, τα ζωικά προϊόντα και ηθική σήμανση και περιβαλλοντική σήμανση. Δεν καταφέραμε να μπουν όλα αυτά στην έκθεση βεβαίως. Αλλά είμαι ικανοποιημένη με τον συμβιβασμό. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την στήριξή μου για αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήθελα όμως να αναφέρω την έλλειψη πληροφοριών σε σχέση με τα χημικά και άλλα προϊόντα για την παραγωγή των υφασμάτων αυτών. Η Κομισιόν μας έχει υποσχεθεί μελέτες από αυτόν και θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για εμάς να λάβουμε αυτές τις μελέτες έτσι ώστε η δημόσια υγεία να είναι πρώτο θέμα. Γιατί βλέπετε πώς εξαπλώνονται οι αλλεργίες. Πρέπει να δούμε τις ε, τυχόν συνδέσεις ε, με αποδείξεις. Σημαντικό είναι να σημειώνονται και τα ζωικά προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για να αυξηθεί η ισχύ του καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι θα αντικαταστήσει αυτό το κείμενο τρεις οδηγίες που είναι ήδη παροχημένες και αφορά τα κλειστοδερικά προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την σήμανση των συστατικών που αποτελούν τα, από τα οποία ε, αποτελούνται τα προϊόντα αυτά. Και η υποχρέωση είναι να αναφέρεται η σύνθεση των προϊόντων. Όμως η απόφαση στο Συμβούλιο είναι αντίθετη από το κείμενο με το οποίο συμφώνησε το Κοινοβούλιο, κυρίως αναφορά το Made in και την ανιχνεσιμότητα των προϊόντων, των κοινωνικών στην ε, σήμανση, στην ετικέτα. Ε, έχει γίνει δεκτή στην Επιτροπή ένα κείμενο το οποίο δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θα καταψηφίσουμε την ε, σύσταση αυτή, διότι δεν δίνουμε τις σωστές πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση και τη σύνθεση των προϊόντων στους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ κύριε Ρώση. Ο κύριος Κόλμαν δεν ε, είναι εδώ, βλέπω καλά. Άρα ακολουθεί ο κύριος Κάντσιεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία, κυρία Υπουργέ για την νέα αυτή νομοθεσία για τα εξωτερικά προϊόντα που θα, υιοθε, που θα υιοθετηθεί αύριο στην Ολομέλεια η Ευρώπη υιοθετεί μια νομοθεσία η οποία δημιουργείται εδώ και χρόνια, έστω και θα αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μια ε, μελλοντική νομοθεσία που θα ολοκληρωθεί αργότερα. Ε, θα πρέπει βέβαια να υιοθετήσουμε κάποια στιγμή και ένα συγκεκριμένο μηχανισμό για την ανεκτευσιμότητα και χαίρομαι γιατί η Κομισιό ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που θα αφορούν τις πληροφορίες που θα αναφέρονται στην ετικέτα και που θα αφορούν την προέλευση και τη σύνθεση των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες και που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές ε, από, τις, από ψευδείς πληροφορίες οι παραπλανητικές πληροφορίες και τον τρόπο αυτό, με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα διευκολυνθούν και οι βιομηχανίες αλλά και οι καταναλωτές διότι θα έχουν και κάποια καινοτόμα προϊόντα και ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα επιβιώσει και θα είναι πιο ανταγωνιστική η θέση της ευρωπαϊκής προστιφετουργίας στην ε, παγκόσμια αγορά θα πρέπει στον τελικό καταναλωτή να δώσουμε μια πιο αληθινή και πιο πλήρη πληροφορία σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία για το Made in και δεν θα επιτρέψουμε οι καταναλωτές να παραπλανώνται. Οι υποχρεώσεις για την επισήμανση για τα κλωστοφωνικά προϊόντα πρέπει να διευρυνθεί και θα πρέπει να προσαρμοστούν ε, οι νομοθεσίες ε, όχι μόνο για τις ίνες και τα κλειστορικά προϊόντα αλλά και, όλοι, και ο κανονισμός για το Made in ε, που υιοθετήθηκε από το, από το Κοινοβούλιο πέρυσι το φθινόπωρο θα πρέπει όσο το πιο γρήγορα να εγκριθεί και από το Συμβούλιο. Ε, κύριε Επίτροπε, μας είπατε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα υποβάλει το κείμενο. Ελπίζουμε ότι όπως μας ε, υποσχεθήκατε θα ε, επιταχύνετε τις διαδικασίε. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Περές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους ε, κατέστησαν εφικτή την επίτευξη συμφωνίας. Μια συμφωνία ε, που πρέπει να μας χαροποιήσει όλους γιατί αφορά την καθημερινή ζωή όλων των ε, πολιτών. Για να είμαι επικοδομητική όπως το συνηθίζω θα ήθελα να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή σας στην σημασία που έχει να δίδονται ακριβείς, εύστοχες πληροφορίες αλλά πάνω απ' όλα κατανοητές πληροφορίες. Να ενημερώνονται οι καταναλωτές λοιπόν για τα συστατικά αποθεματικά των κλωστεφαντορικών προϊόντων. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα πλήρη και εξωτερική ενημέρωση, αν δεν μπορούν ε, όμω να την αποκωδικοποιήσουν όλοι οι συμπολίτε μα. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ θετικό βήμα, αλλά δεν είναι επαρκέ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να προστατεύσουμε του πολίτε ε, που θα μπορούσαν να είναι και οι πλέον ευάλωτοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίε και κύριοι, να θεσπίσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, σήμανσης και των μεγεθών με βάση σωματικέ διαστάσει, ώστε όταν πάμε να αγοράσουμε ένα ε, ρούχο όπω τώρα να προσέχουμε το, το μέγεθος, γιατί αυτό είναι το βασικό που κοιτάμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αναρμόνιση στα μέγεθα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κύριος Σμιτ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μάντερς. Χαίρομαι για το ότι συμπεριλαμβάνεται τώρα και η πτυχή της υγείας και το θέμα της γούνας. Ξέρουμε πως είναι σημαντική η σήμανση και η επιλογή του καταναλωτή και αν είναι να επιλέξουν σωστά οι καταναλωτές χρειάζονται πληροφορίες εύληπτες και αξιόπιστες. Σήμερα λοιπόν έχουμε ρούχα με υλικά από πάρα πολλές χώρες οπότε είναι αδύνατο να πούμε που έχουν κατασκευαστεί. Τα ανέφερε και ο κύριος Μάντερς. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα πούμε. Πώς θα πούμε ποιο κομμάτι είναι από ποια χώρα. Ξέρετε πως η προέλευση σε αυτό τον κόσμο το παγκόσμιο είναι ένα μέσο καλύτερης ε, πληροφόρησης αλλά μπορεί να είναι και ένας αντιπερισπασμός προστατευτισμού. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο και ε, αυτό έχει κάνει την Ευρώπη μεγάλη. Ευχαριστώ κυρία Ρόσμπαχ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο τομέας αυτός είναι παγκόσμιος, ε, τα ρούχα συχνά κάνουν το γύρο του κόσμου μέχρι να γίνουν τελικό προϊόν. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυτεχνική έκθεση και βρίσκει τη δύσκολη ισορροπία μεταξύ του δικαίωματο, πληροφόρηση των καταναλωτών, λασιμότητα και ανταγωνιστικότητας. Οι καταναλωτέ έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες χημικέ ουσίε ε, περιλαμβάνονται στην κατασκευή του προϊόντος, από πού έχει έρθει το προϊόν και τα Αλλά τι γίνεται ε, με την ισορροπία ε, και μια απλή ετικέτα που γράφει οδηγίες πλησίματος και τη διαφορά με ένα τεράστιο πάπυρο που θα γράφει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε. Ο συμβιβασμός αυτός λοιπόν πηγαίνει σωστή κατεύθυνση αλλά θα ισχύσει μόνο το 2013 που θα έχουμε και τα αποτελέσματα της Κομισιόν και άρα θα έχουμε ένα πλαίσιο για το πώς οι καταναλωτές θα μπορούν να έχουν ακριβείς πληροφορίες για πώς θα έχουμε και πλήρη χνηλασιμότητα της παραγωγής φασμάτων και ελπίζω έτσι να οδηγηθούμε σε λογική νομοθεσία μέχρι το 2013 οπότε ελπίζω και χαίρομαι για το ότι η Κομισιόν θέλει να φέρει πιο νωρίς την ημερομηνία εφαρμογή. Ευχαριστώ κυρία Ρόσμπαχ για ένα λεπτό ένα Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το 2005 η κατάργηση των κλωστογενικών ποσοστώσεων άνοιξε τις πόρτες της ε, Ευρώπης στο ντάμπινγκ και αυτό ήταν ε, πολύ καταστροφικό και για την οικονομία και για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία των καταναλωτών μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, υγεία των καταναλωτών, την υγεία των εργαζομένων στο τομέα και υπό, έστω και αν δεν προχωράνε πάρα πολύ υποστηρίζουμε τις προτάσεις που γίνονται όσον αφορά ε, ε, τις, την παρουσία επιβλαβών ουσιών, την σήμανση των προϊόντων. Θα πρέπει όμως οι πληροφορίες αυτές να εμφανίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη και να, τον, ε, την παραχάραξη, την παραποίηση των προϊόντων να την πατάξουμε σε όλες τις χώρες. Είναι θέμα πολιτικής θέλησης. Θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι δεν μας, ενδιαφέρουν, ε, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, τόσο πολύ τα πλαστά, το πλαστό προϊόν όσο και η, ε, το να σταματήσουμε τους λαθρομετανάστες στα σύνορα Ιταλίας-Γερμανίας, ε, Ιταλίας-Γαλλίας. Ευχαριστώ. Επίσης για ένα λεπτό, κύριο Σαλβίνη. Grazie Presidente. Io voglio Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο Ταγιάννη για την ε, προσπάθεια. Πρέπει να σας πω ότι είναι σουρεαλιστική συζήτηση, διότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Μας κοροϊδεύουν εδώ. Άκουσα κάποιον αριστερό, κάποιο συνάδελφο της αριστεράς ε, να ζητοκραυγάζει. Εμείς όμως δεν ξέρουμε από πού προέρχονται τα προϊόντα τα οποία φοράνε οι καταναλωτές. Υπάρχει το ελεύθερο εμπόριο. και, υπάρχει και η φωνή το κάποιων εμπόρων που έχουν ε, επιζήσει ε, καταλαβαίνω βέβαια ότι θα πρέπει να γίνει ένα συμβιβασμό. Το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε μέσα στα πλαίσια της πρώτης ανάγνησης ήταν ένα καλό ε, κείμενο το οποίο προστάτευε τους καταναλωτές και τους ε, κατασκευαστές. Μετά όμως έγινε μια καταστροφή. Κανείς δεν ξέρει ε, τι φοράει ο καταναλωτής ε, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει το Συμβούλιο ή την φωνή των ε, καταναλωτών δεν την ακούει το, δεν την άκουσε η Ουγγρική Προεδρία φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακριά από τους πολίτες της Ευχαριστώ για δύο λεπτά ο κύριος Σάγκεντη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Αντιπρόεδρε. Επιτρέψατε μου να αναφέρω δύο σημαντικά ζητήματα εδώ πέρα. Πρώτον, πώς είναι σημαντικό στην ετικέτα να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. Και δεύτερον, η ουσία από την οποία αποτελείται το προϊόν. Και καλό είναι να έχουμε και για τις δύο περιπτώσεις ενιαίους κανόνες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, για το ζήτημα της κατασκευής και προελεύσεως. Ε, υποθέτοντας ε, και όλας βεβαίως πως υπάρχει μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το δεχόμαστε, και πως πάρα πολλοί κλάδοι όπως και η κλωστοϊφαντουργία ε, πλήττονται από τη μετατόπιση της παραγωγής σε άλλες χώρες, στην Ασία δηλαδή. Οπότε θα πρέπει να βρούμε δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και στον τομέα της κλαιστοϊφαντουργίας, μηχανουργίας, γεωργίας, τουρισμού, όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν ότι αντιμετωπίζουν κρίση. Η ευρωπαϊκή παραγωγή έχουν και μειονέκτημα με όλα αυτά τα φτηνά προϊόντα, προϊόντα dumping από την Άπο Ανατολή που καθιστούν σχεδόν αδύνατο τον ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Και ίσως θα έπρεπε και κατασκευαστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναφέρονται στην ετικέτα για να βλέπουν οι καταναλωτές στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και την Τσεχία εάν θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί και στη χώρα τους. Σημαντικό είναι να ξέρουμε επίσης την ποιότητα των ινών και αυτό βέβαια θα το κρίνουν τα εργαστήρια. Σας ευχαριστώ κυρία Ρόιτοβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχει περάσει περίπου ένας ε, χρόνος, παρά μια εβδομάδα, από τότε που μια μεγάλη πλειοψηφία είχε υπερψηφίσει μια πολύ ε, συνολική πρόταση της Επιτροπής ΙΜΚΟ στην πρώτη ανάγνωση για τη σήμανση των κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Για εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά του κύριου Μάντρης και των υπολείπων που μέχρι τελευταία στιγμή προσπάθησαν με το Συμβούλιο να διαπραγματευτούν μια κοινή θέση σε δεύτερη ανάγνωση, ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην παραγωγή ταχύτερα νέε φάνσιμε ίνε, αλλά και να βελτιωθεί ασφάλεια. Λυπούμε όμως, αλλά το Συμβούλιο επιμένει και αρνείται την εναρμόνιση των μεγεθών και τη σήμαση της χώρας προέλευσης. Ε, ε, αρνείται έτσι στους καταναλωτές το δικαίωμα να γνωρίζουν που έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος το οποίο αγοράζουν. Ε, δεν μιλάμε για μυστικά εδώ πέρα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και αν ε, πρέπει να, και, και, πρέπει να είναι υπερήφανοι οι καταναλωτές μας για τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε, σε χώρες με φθηνό δυναμικό. Πρέπει να υπάρξουν καλύτεροι έλεγχοι παρά τους οποίους εισέρχονται πάρα πολλά προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να γίνει επίσης μια μελέτη επιπτώσεων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, η οποία όμως να επικεντρώνεται όχι μόνο στη χώρα προέλευση, αλλά και στις εναρμονισμένες μεθόδους κατεργασίας, στα μεγέθη, στο κατά πόσο περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, αν είναι έφλεκτα κτλ. τα προϊόντα. Πρέπει ε, να μην προασπίζει η Κομισιόν περισσότερο τα συμφέροντα των εμπόρων και λιγότερο αυτά των πολιτών και των καταναλωτών. Και ε, το πώς και πώς θα μπορέσει να αλλάξει το Συμβούλιο άποψη δεν ξέρω, αλλά πρέπει ε, και εδώ ε, αλλά και στις χώρες μας ο καθένας να συζητά με τις κυβερνήσεις να προσπαθεί να τις μεταπίσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο μάντρη, αλλά και όλους για, για το σημερινό επίτευγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σούστα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση κανονισμού θα πρέπει να μας βρει σύμφωνους, διότι ε, διευκολύνει και τα κράτη-μέλη. Και ε, συμφωνώ με, τις, ε, με την Επιτροπή όσον αφορά την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών του εξωτερικό τομέα. Ο κανονισμός αυτός ε, διευκολύνει και την διαφάνεια, διευκολύνει την ε, πώληση των προϊόντων αυτών. Βέβαια, η ρήτρα επανεξέτασης ε, και ο συμβιβασμός με το Συμβούλιο για την προέλευση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα προηγούμενο και, θα, και να θέσει θα αποδυναμώσει την θέση, θα αποδυναμώσει την διαπραγμάτευση ανάμεσα στο, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και στο, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη την δημοκρατική φωνή που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λάβει υπόψη τις απόψεις των βουλευτών. Ε, βέβαια, εμείς θα υπερψηφίσουμε το, το κείμενο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό, κύριος Μορκαντή. Πρόεδρε, ο κανονισμός αυτός ε, έχει πολύ χρήσιμες διατάξεις, ε, διότι διευκολύνει τα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν καταφέραμε να εντάξουμε στον κείμενο και μία αναφορά στο σήμα προέλευσης. Για τον κλειστορικό τομέα αυτή η διάταξη θα ήταν ε, ουσιαστική σημασία και θα ήταν μία εγγύηση και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Οι βασικοί μας ανταγωνιστές, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία και η Κίνα εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό την ίδια ρήτρα για τα εισαγόμενα προϊόντα. Η Ευρώπη, και δεν καταλαβαίνω κανένα το λόγο, θεωρεί ότι το θέμα αυτό είναι άσχετο και περιττό. Όμω, επί του παρόντο, ε, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, διότι μια τέτοια ε, ετικέτα, εκτό από την προστασία και την εγγύηση τη ασφάλεια, θα μα διευκολύνει για την, να, να, να πατάξουμε και την, ε, τα πλαστά. Στο Πράτο, πριν από λίγο καιρό, στην χώρα, στην πόλη μου δηλαδή, βρήκαμε με ένα μεγάλο αριθμό πλαστών προϊόντων που προέρχονταν από την Άπο Ανατολή και ήταν ε, πάρα πολύ φτηνά. Η Ευρωπαϊκή κλειστοεφαντουργία έχει γονατίσει και πιστεύω ότι ούτως ή άλλως κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Κυρία Κόμι, είχατε ένα ερώτημα προς ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους ε, από την ε, Λέγκα του Βορρά τι έκανε ε, το κόμμα, κόμμα σας στον τριμερή διάλογο γιατί ζητήσαμε να συνεισφέρετε ενεργά. Εγώ το ζήτησα και το ΕΛΚ. Εγώ και το ΕΛΚ το ζητήσαμε. Επομένως είναι εύκολο να κριτικάρει κανείς αλλά θα πρέπει πρώτα όμως να συνεργαστεί με τους άλλους. Λέτε να απαντήσετε. Στην πρώτη, ανάγνωση ε, στην Επιτροπή είχαμε ένα άλλο κείμενο και εκεί υπήρχε το πιστοποιητικό προέλευσης του προϊόντος και δεν καταλαβαίνουμε γιατί το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό, στο Συμβούλιο και η Κομισιό υποχώρησε. Εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε. Επομένως το κείμενο αυτό εμείς δεν θα το υπερψηφίσουμε λόγω ακριβώς ναι, του ότι δεν υπάρχει το, ε, η πιστοποίηση προέλευσης. Ο κύριος για δύ- η κυρία Γκαρδίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι όλοι εδώ προσπαθούμε να αξιολογήσουμε ένα κείμενο το οποίο έχει κάποια κενά βέβαια. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε ένα κείμενο πιο φιλόδοξο όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά επίσης όλοι συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Είναι προφανές ότι ένα σαφές υποχρεωτικό σύστημα για την ετικετοθεσία επιτρέπει ένα καλύτερο έλεγχο, επιτρέπει να πατάξουμε τις απάτες, ε, διασφαλίζει την νομιμότητα κτλ. Και όλοι χαιρετήσαμε το γεγονός ότι με το κείμενο αυτό εντάσσεται η υποχρέωση ε, ε σήμανσης ε, των ε, στοιχείων που δεν είναι, ε, που είναι ζωικής προέλευσης και είναι το κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στην αγορά Μάλλον προσπαθούμε να αποτρέψουμε την παρουσία στην αγορά μας στοιχείων στα προϊόντα, τα γούνας παραδείγματος χάρη που προέρχεται από σκύλους, γάτες κτλ. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε κανόνες προστασίας του καταναλωτή, του εργαζόμενου, του περιβάλλοντος, του ανήλικου, ε, θέματα που θεωρούνται δεδομένα στην Ευρώπη και που ε, αποτελούν μια εγγύηση για τους πολίτες μας και τους καταναλωτές. Όλοι πρέπει να γνωρίσουμε ότι ε, πρόκειται για μια μάχη την οποία θα πρέπει να νικήσουμε μαζί όλοι μαζί. Είναι ένας αγώνας τον οποίο δίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εδώ τώρα έχουμε κερδίσει μια σημαντική μάχη στον πόλεμο αυτό. Αυτό το οποίο ε, ανέλαβε να κάνει ο, ο Επίτροπος είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το κλειστοδικό το τομέα, αλλά για όλους τους τομείς, ε, διότι πιστεύουμε ότι ο καταναλωτής ε, πρέπει να ξέρει ποια είναι η χώρα προέλευσης. Είναι το βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει και θέλει να ξέρει ο καταναλωτή. Και πιστεύω ότι ε, είναι ένα κείμενο πάρα πολύ σημαντικό. Σα ευχαριστώ κυρία Γκαρδίνη. Περνάμε στη διαδικασία ε, και και θα δώσω τον ε, λόγο στην κυρία Κάλπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πέρα βεβαίω μιλάμε για τα συμφέροντα των καταναλωτών και θα πρέπει να είναι και κατανοητές οι ετικέτες. Γιατί στις ετικέτες ε, στηριζόμαστε για να έχει την ενημέρωση και την προσθέμενη αξία ο καταναλωτής. Βεβαίως η κατάσταση αυτή ε, η σημερινή σημαίνει ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επανεξετάζουμε νομοθεσίες οι οποίες δεν θα είναι πλέον επίκαιρες. Τώρα για το θέμα επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο επισταμμένος. Να δούμε αν υπάρχει πράγματι αιτιώδης ε, σχέση μεταξύ χημικών, συνθετικών ουσιών και αλλεργικών αντιδράσεων. Θα πρέπει να επιμείνουμε άρα πολύ περισσότερο στην ποιότητα στο μέλλον και βεβαίως η χνηλασιμότητα παίζει εδώ πέρα ρόλο. Ευχαριστώ κυρία Γκάλ Πέλτς και τελειώσαμε με αυτή τη διαδικασία. Να δώσω τον λόγο λοιπόν στην κυρία Πρέντεργας. Μικρόφωνο κυρία συνάδελφε. Τώρα το άνοιξα. Ευχαριστώ. πολίτες τη Ένωση έχουν δικαίωμα να ξέρουν την σύνθεση των προϊόντων και των ρούχων που φοράνε και τώρα θα ξέρουν αν έχουν κομμάτια ζωικής προέλευσης για λόγους υγείας, ηθικής ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα οποία θεωρούμε π.χ. ω γιακάδε, στολίδια κτλ. δεν ε, αναγράφονται υποχρεωτικά στην σήμανση. Ήδη υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετική για τα παπούτσια και λογικό είναι να υπάρχει και για τα ρούχα. Ειδικά όσοι έχουν αλλεργίες θα υποφεληθούν από αυτή την πρόταση, καθώς μπορεί να υπάρχουν ουσίες ε, πιθανώς ε, βλαβερές για την υγεία και η Κομισιόν πρέπει να δει τις σχέσεις μεταξύ ε, επικίνδυνων χημικών ουσιών και αλλεργικών αντιδράσεων και θα πρέπει στο μέλλον να δούμε τα επιστημονικά δεδομένα για τις αλληλικές αντιδράσεις και βεβαίως πρόκειται για ισορροπημένες προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρέντεργκαστ. Να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση τεχνικού χαρακτήρα, αλλά είναι μια συζήτηση πολιτικού χαρακτήρα που εντάσσεται στην, στο πλαίσιο των επιλογών που πρέπει να κάνουμε για την πραγματική οικονομία από πλευράς των ευρωπαϊκών θεσμών, από το Κοινοβούλιο, από το, την Κομισιό και το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Επίτροπος θέλει να προστατεύσει την πολιτική της βιομηχανίας, την, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δώσουμε μια εγγύηση και στους καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων μας. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετράται επίσης και από την ποιότητα των προϊόντων όταν έχουμε να κάνουμε και με την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα το βράδυ, στο τέλος αυτής της συζήτησης, επαναλαμβάνει την θέλησή της να προχωρήσει όσον αφορά την υλοποίηση του Made in. Ε, θα επιταχύνουμε τις ε, διαδικασίες και τις προθεσμίες. Θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο Καντσάν αλλά και τους άλλους ε, βουλευτές που είπαν ότι οι προθεσμίες είναι μεγάλες κτλ. Όπως είπα και στην αρχική, του, στην αρχική μου ομιλία έχω ήδη δώσει εντολές στις υπηρεσίες μου να προχωρήσουν, να συνεχίσουν στο δρόμο που ξεκινήσαμε, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν στο πλευρό του Made in, υποστήριζε το Made in και για τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όσον αφορά τα προϊόντα τα εισαγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνω μια έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το Συμβούλιο μάλλον σήμερα, γιατί η συζήτηση δεν ήταν τόσο καρποφόρα. η κυρία Γιώρη μας είπε ότι το Συμβούλιο δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ρήτρα την οποία, για την οποία συζητάμε που αποτελεί και το κλειδί για την πολιτική συζήτηση. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να βρει μια λύση, όχι υπαναχωρώντας, αλλά προχωρώντας, έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στους καταναλωτές. Το θέμα της ανεκτευσιμότητας αφορά και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ήταν η πρωταρχική μου ε, προτεραιότητα από την αρχή όταν ξεκίνησα σαν επίτροπος να προστατεύω τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, συνεχίζω στηρίζοντας ε, το έργο του προκατόχου μου και έτσι θα συνεχίσω να προφυλάσω και να προστατεύω την ε, ε, υγεία των καταναλωτών, διασφαλίζοντας όμως και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία πρέπει να είναι ε, Στι πρώτε θέσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι η ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία εξαρτάται από την ποιότητα. Γι' αυτό θέλω να συνεχίσουμε τι εργασίες. Εγώ είμαι ικανοποιημένο από τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ανάμεσα στου σύνομοθέτε, αν θέλετε, γιατί ξέρετε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι οι νομοθέτε που θα ε, ολοκληρώσουν το κείμενο στη δεύτερη ανάγνωση. Αλλά και εμεί, σαν Επιτροπή θέλουμε από να συνεχίσουμε το έργο έτσι, το, και την, ε, τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, να διασφαλίσουμε τα γνωστικότητα των προϊόντων μας. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω και την, ε, υπό, τις, δεσμεύσεις μας για να προωθήσουμε την ε, καινοτομία στον τομέα των κλωστοϊδουργικών. Η βιομηχανική, η πολιτική βιομηχανική έχει στα σκαριά πολλά πράγματα ακόμα. Ε, και θέλουμε να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στην ε, βιομηχανία και να συγκεκριμενοποιήσουμε την παραγωγή νέων προϊόντων ε, διότι αυτό αποτελεί και ένα σημαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της μόδας. Διότι η βιομηχανία μας τι είναι, είναι ανάπτυξη και είναι και θέσεις απασχόλησης, ε, είναι η θέση μας στην αγορά. Ε, η αγορά δεν έχει βέβαια κανένα νόημα εάν δεν ε, λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική πτυχή. Αν δεν υπάρχει πολιτική, κοινωνική πολιτική, τι δεν κάνουμε την αγορά. Σας ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στην κυρία Γκιόρη, εξ του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Θα αναφερθώ σύντομα στις παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά την ένδειξη προέλευσης. Ήταν και το συναρπαστικότερο τμήμα. Όχι μόνο στις διαβουλεύσεις, αλλά και εντός του Συμβουλίου ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Επειδή στον τομέα της εμπορικής πολιτικής δεν είχαμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τις οριζόντιες διαβουλεύσεις. Δεν θεώρησα σωστό να δημιουργήσω κάποιο προηγούμενο εδώ πέρα με το να δημοσιεύσουμε κάτι πάρα πολύ νωρίς. Είδαμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά την προέλευση και την σήμανση τη σχετική Αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν ήδη σε εθελοντική βάση. Αν όμως ε, τηρήσουμε κάποια κριτήρια θα οδηγηθούμε σε κάποιες ε, στρεβλόσκα, κάτι το οποίο βεβαίως θα θέλαμε. Είμαι σίγουρη πως η Κομισιόν θα ε, μελετήσει τυχόν επιπτώσεις ενός τέτοιου συστήματος. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Επίτροπο Ταγιάννη για την δέσμευση την οποία ανέλαβε να επιταχύνει τις διαδικασίες στην Κομισιό έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη τόσο σημαντική υπόθεση. Ε... Και αυτό αποφασίσαμε την εξή λύση, μια ρήτρα αναθεώρησης και μια αιτιολογική σκέψη και χαρήκαμε για το ότι η κυρία Λάρα Κόμη, η οποία βεβαίως είναι και ε, η σημαντικότερη αντίπαλος του θέματος αυτού, θεωρεί το ζήτημα αυτό και τη λύση αυτή ικανοποιητική. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχουμε τώρα ε, για το μέλλον ε, μια πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απάτη και σημαντικό είναι να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδες ηγητές, βουλευτές της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Γκέρη. Τον λόγο έχει πάλι ο κύριος Μάντερς για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε πως η Επιτροπή μας είναι πάντα υπέρ του ελευθέρου εμπορίου και κατά του προστατευτισμού. Ποτέ αυτό δεν θέλαμε. Εμείς θέλαμε να ε, υπάρχει ενημέρωση του ε, καταναλωτή. Και έχω βαρεθεί να ακούω τους ε, συναδέλφους που λένε πως περάσαμε κάτι στη, με το να μην συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση κτλ. Μα αν δεν θέλει η Κομισιόν και το Συμβούλιο δεν περνάμε τίποτα. Και είδα τον κύριο Ταγιάννη ε, πόσο στήριξε τον συμβιβασμό μας και ελπίζω κυρία Υπουργέ, κυρία Γκέρι, να μπορέσετε να πείσετε το Συμβούλιο να αναδεχτεί τα θετικά <coughs> αποτελέσματα της μελέτης. Και αν γίνει κάτι τέτοιο θα δείτε πώς θα έχουμε κατα... νομοθεσία καλή για τον καταναλωτή και την βιομηχανία γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε ενδύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ και τον κύριο Ταγιάννη για τη στήριξη και ελπίζω να έχουμε σύντομα τα αποτελέσματα της έρευνας και η Προεδρία του Συμβουλίου να πείσει το Συμβούλιο να αποδεχτεί αυτά τα αποτελέσματα. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε πως το μέλλον θα αποδείξει πως ε, έχουμε εδώ πέρα ένα πρότυπο για πάρα πολλούς τομείς Δηλαδή να μην ε, έχουμε νομοθεσία η οποία ε, δεν θα στηρίζεται, αλλά θα έχουμε μια νομοθεσία η οποία θα στηρίζεται σε επιστημονικά επιχειρήματα με συνεισφορά όλων των, των συναδέλφων και άρα θα είναι και περισσότερο αποδεκτή από όλους στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μάντερς. Τελειώνει άρα η συζήτηση. Η ισοφορία θα γίνει αύριο στις 12.30 ώρα. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, προφορικές ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή που αφορούν τα τεστ